ολοκληρωτισμό στην ιστορία της χώρας του. Λοιπόν, εδώ λίγη η συνεδρίαση της Ολομέλειας. Ε, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας για αυτή τη Σύνοδο Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια συζήτηση που ήταν ε, πιο ε,